Der Präsident! Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Επαναλαμβάνεται οι συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτο σημείο της ημέρησης διάταξης είναι η έκθεση Μπαχ για τις αποζημιώσεις για τους επιβάτες αεροπορικών εταιριών και η παροχή βοήθεια σε αυτούς σε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησης επιβίβασης ή ματέωσης μιας πτήσης και δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Μπαχ.